Αγαπητοί συνάδελφοι, ακολουθεί η ψηφοφορία. Έκθεση του κυρίου Σπερώνη πρώτα, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα θέλει και το λόγο. Ναι. Apparently not. Α, όχι. Καλώς τότε. Α, θέλει. Me? Therefore, I will put the report... Τότε να ψηφίσουμε. Ο κύριος Γκολνής θέλει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, το γνωρίζετε, διότι και εσάς την ίδια σας έδωσε άδικο ε, σε το ΔΕΚ, σε ένα θέμα που με αφορά και ελπίζω η επίοικια που επιδεικνύεται απέναντι στον κύριο Μπρόκ για ένα θέμα οικονομικό να ισχύει και σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφραση των βουλευτών του Κοινοβουλίου που είναι στη μειοψηφία. Αυτή η ισότητα που επικρατούσε πριν από 20 χρόνια στο Κοινοβούλιο ε, το τιμούσε και τιμούσε και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δυστυχώ, το θέμα των ασυλιών άλλαξε με τρόπο μέρο λυπτικό και λυπάμαι γι' αυτό και ελπίζω να συνέλθει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. We will now move... Προχωρούμε στην ψηφοφορία της έκθεσης κυρίου Σπερώνη. Α, ο κύριος Σπερώνη θέλει το λόγο, ο οποίος ήρθε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα δει ε, ότι η ψηφοφορία άρχιζε στις 12.25. Ε, το μόνο που θα ήθελα να διευκρινίσω είναι ένα αριθμητικό στοιχείο. Εκ παραδρομής στις αιτιολογικές σκέψεις γίνεται λόγος για 2.900 ευρώ, ενώ το ποσό είναι 2.356,41 ευρώ. Αυτό. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση αυτή και τώρα ψηφίζουμε. Παρακαλώ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε Σπερώνη. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση της κυρίας Σάλντε Μόζε, Γενική Ασφάλεια Προϊόντων και Εποπτεία της Αγοράς. Είναι μία ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Συγχαρητήρια ε, προς την εισηγήτρια. Επόμενο θέμα η ψήφιση τη έκθεση κυρία Ριβαζή, διαχείριση της γρήπης ΙΤΑ 1 1 και πάλι μία ε, ψηφοφορία ψήφι κατά εποχέ εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά και πάλι συγχαρητήρια κυρία Ριβαζή. Επόμενο θέμα. Ο διορισμός μέλους του Ελεκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι για τον κύριο Χάραντ Βέγγερ Μπάουερ, έκθεση τη κυρία Σαγιάλα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεν θα δείτε το αποτέλεσμα, ένα γαλάζιο φως θα δείτε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται και ο διορισμός αυτός. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Επόμενο θέμα. Ε, έκθεση Ριβελίνη περιοχή της Συμφωνίας Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο. Πρόταση κανονισμού. 39 τροπολογίες Επιτροπής Αλίας ψηφιπέ κατά απόχες εγκρίνεται. Το σύνολο των τροπολογιών αυτών. Τροπολογία 41 με ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι Κατά αποχές Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 48 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 49 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 50 ψήφι π. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 51 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 52 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 47 ψήφι π κατά αποχές εγκρίνεται και η 12 α, συγγνώμη, διορθώνει Πρόεδρος το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ονομαστική κλίση α, κάτι ξέχασα η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε ψηφίπε. κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Everybody Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον σύγητη. Και τώρα ερχόμαστε στην έκθεση της κυρίας Ποδηματά με θέμα την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γκοζές πριν ψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 1. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτής της κυρίας Ποδηματά ε, γίνεται λόγος για σημαντικά ζητήματα για την καινοτόμο χρηματοδότηση και λυπάμαι γιατί έχει προκληθεί κάποια σύγχυση και θα παρακαλούσα την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να αποσύρουν το εναλλακτικό ψήφισμα που πρότειναν ε, έτσι ώστε ε, να ε, έρθει σε έσω πέρα η κοινή προσπάθεια και το προϊόν αυτής. Λυπάμαι που στο θέμα του τέλους των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχουμε δύο τροπολογίες πάρα πολύ όμοιες μεταξύ τους. Λυπάμαι, γιατί έτσι δεν θα ε, μπορέσει το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει μαζικά αυτό το τέλος ε, σε όρους ε, φρονιμότητας και σοφροσύνης σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ. Κύριο Σούλτς, από ό,τι κατάλαβα, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να πω στον συνάδελφο Γκοζές ότι αυτό το σχέδιο εναλλακτικού ψηφίσματος μάλιστα θα το αποσύρουμε. Συνέστησα στην ομάδα μου να το κάνει για τον εξή απλούστατο λόγο. Η επόμενη τροπολογία που έχουν υποβάλει 120 συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες δείχνει το εξής, ότι το θέμα του τέλους των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν είναι πρώτα σοσιαλιστική ή του ΕΛΚ ή των Πρασίνων ή των Συντηρητικών, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε μια θεσμική πρόταση, να δώσουμε ένα θεσμικό μήνυμα το Κοινοβούλιο εδώ πέρα από πολιτικές ομάδες να πούμε ότι είναι σε θέση να πει ότι ο τομέας της ιδιωτικής οικονομίας θα πρέπει να αναλάβει το μερίδιο που του αναλογεί στην καταπολέμηση της κρίσης. Αυτό δεν είναι σοσιαλιστικό, δεν είναι συντηρητικό, είναι κοινή μας βούληση. Αν θέλουμε να την εκφράσουμε σήμερα θεσμικά, αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό και αποσύρουμε την λόγο τροπολογία. Πρόεδρε, χθε στην Ολομέλεια κάναμε και μια άλλη πρόταση από την μεριά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, αν μπορεί να γίνει σαφέ και θα μπορούσε να είναι ένα συμβιβασμό, ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν στον κοινοτικό προπολογισμό και στο μηχανισμό στήριξη. Θέσαμε το θέμα στην, ε, συζήτηση εχθέ και περιμένουμε την απάντηση για να κάνουμε ένα συμβιβασμό και ένα θετικό μήνυμα να στείλουμε προς το, στα κοινοτικά όργανα. Ευχαριστώ. Uh, Κοιτάξτε, βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία τώρα. Αποσύρθηκε η πρόταση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες τροπολογίες όπως έχουν προβλεφθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε μέσω τώρα στην τροπολογία παριθμών 2 με ονομαστική κλίση ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία παριθμών 2. Άρχεται τώρα η ψηφοφορία. Να ψηφίσετε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα προχωρούμε στις μεμορωμένες παραγράφους. Η παράγραφος 20 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 32 σε ψηφοφορία κατά τμήματα και τα δύο ονομαστικά. Το πρώτο τμήμα της 32 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 32 αρχίζει ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται επίσης. Η παράγραφος 36, ψήφιπε Κατά, αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 39, ψήφι Κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 40. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ γιατί 40 γιατί δεν ήταν σαφές. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, παράγραφο 42 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λέει η πρόεδρο, αλλά στο ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά για τη 42. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Όχι, απορρίπτεται. Η παράγραφος 65 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Το σχέδιο ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγητριά μας. Το επόμενο σημείο είναι η ψηφοφορία της έκθεσης Εστρέλα με θέμα τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Η κυρία Άουγκεν ζήτησε το λόγο. Ε, er Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τους Δανούς. Στη δανική μετάφραση η λέξη equitable έχει μεταφραστεί λάθος γιατί ε, ε, πρέπει να αλλάξει. Είναι ένα θέμα γλωσσικό ε, και δεν ξέρω αν έχουν το ίδιο πρόβλημα οι Σουηδοί. Αντί για ίσο πρέπει να είναι ισότιμο. Είναι ένα θέμα μετάφραση, σε πάση περιπτώσει, τη έκθεση στα δανεικά. Σα ευχαριστούμε, κύριε Άουκεν. Ψηφίζουμε. Παράγραφος 4. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Δύο τμήματα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Oh, sorry, the first part not with Συγγνώμη, όχι ονομαστικά το πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Σε δύο τμήματα. μάλλον σε τρία τμήματα παράγραφος 5. I've been given the wrong λάθος κείμενο μου έχουν δώσει. Για το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπερχωρής ονομαστική ψηφοφορία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσετε, τέλος. εγκρίνεται και τρίτο τμήμα της παραγράφου 5 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία έχετε ψηφίσει όλοι ναι τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται παράγραφος 6 Ψηφοφορία σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Τέλος. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα και τώρα το δεύτερο τμήμα χωρίς ονομαστική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το παράγραφος 7. Παράγραφος 8 δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Είμαι μάλλον λάθο. Το πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. And Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. Παράγραφος 22. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 25 σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 25. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Σε δύο τμήματα. Άρχεται ψηφοφορία ονομαστικά για το πρώτο τμήμα. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 29. Τέλος. Αυτό απορρίπτεται. Παράγραφος 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 37. Σε δύο τμήματα ποιος είναι υπέρ του πρώτου. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, εντάξει, ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 37. Τέλος. Εγκρίνεται όντως. Παράγραφος 53 σε δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία μόνο για το δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου καταρχήν. Κατά αποχές. Οριακή διαφορά. Θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 53. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση για την παράγραφο 53. Δεύτερο τμήμα, αρχή ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 56. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 57 σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική κλίση για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 57. Έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 64. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 77, ε, παράγραφος 76, παράγραφος 77 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Δέλτα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, G με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται η αιτιολογική σκέψη G. Ε, αιτιολογική σκέψη H με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Άι, με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Ε, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη O, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 2α σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ κατά, οχές. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α δέλτα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος, εγκρίνεται. Τώρα το σχέδιο ψηφίσματος ολόκληρο άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Συγγεντρία. και περνάμε στην έκθεση Εύας Ζολή, συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, παράγραφος 10, σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, οριακή διαφορά. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την παράγραφο 12 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καλώ σας στείλουμε τεχνικό. Παράγραφο 15, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα τη παραγράφου 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι οριακή διαφορά. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την παράγραφο 19. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33 και πάλι σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 33. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλώ, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πολύ ευχαρίστω. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1 παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 39. Σε τρία τμήματα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 39. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα της παραγράφου 39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 43. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 66. Σε δύο τμήματα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 68. Σε δύο τμήματα, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Οριακό το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την αιτιολογική σκέψη G. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, λέει η Πρόεδρος. It is the original text. Πρόκειται για το αρχικό κείμενο, άρα σε περίπτωση ισοπαλίας εγκρίνεται όταν η τροπολογία πάλι οδηγεί στην απόρριψη. Είναι το αρχικό κείμενο. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη H. Ποιο είναι υπέρ. Those against. Κατά αποχές. Ασαφές το αποτέλεσμα. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την αιτιολογική σκέψη H. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, λέει η Πρόεδρος. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Λάθος, διορθώνει η Πρόεδρος. So the motion... Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση είναι του κυρίου Παπαστάμκου για τη γεωργία και το διεθνές εμπόριο. Παράγραφος 3. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απόχέ. αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος αφού επιμένετε, γιατί μερικοί δεν σήκωναν τα χέρια. Εν πάση περιπτώσει, δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονικός έλεγχος για την παραγραφό 12, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ασαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για το τρίτο τμήμα της παραγράφου 12. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 13. Σε δύο τμήματα, ποιος είναι υπέρ του πρώτου, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 και πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Voted, voted. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21 σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 43 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. You've all voted. Vote is Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 45 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 47. Σε 7 τμήματα. Ελπίζω να με βοηθήσετε στο μέτρημα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματο. Κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πέμπτο τμήμα της παραγράφου 47. Voted, the vote is... Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. And that is adopted. So we now... Εγκρίνεται. Έκτο τμήμα 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι ήταν οριακή διαφορά. Έλεγχος και για το έκτο τμήμα της παραγράφου 47. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στο έβδομο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 48 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 49 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 49. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 51 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 52 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 53. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 53 ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 53. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 54. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 59. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη R. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο του νομοθετικού ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. The next item Επόμενη η έκθεση του κυρίου Χόισλινγκ, το πρωτοεινικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 80% πρωτεϊνικό έλλειμμα έχει η Ευρώπη και θα πρέπει να μειωθεί με ε, υποστήριξη της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, στην έκθεση δεν ε, είναι θέμα να γίνει συζήτηση για τη μηδενική ανοχή ή πώς θα διευκολύνεται η εισαγωγή γενετικά τροποποιημένης τροποποιημενη σογιας Γι' αυτό παρακαλώ να καταψηφίσετε την έκθεση 3 και, τη, συγγνώμη, την τροπολογία 3 και 9, διότι αν εγκριθούν αυτές οι τροπολογίες, αλλοιώνεται τελείως η έκθεση και θα υποχρεωθώ να αποσύρω το όνομά μου. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στη ψηφοφορία. Ε, παράγραφος 2 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. And that is adopted. Paragraphs... Εγκρίνεται. Παράγραφος 3 και πάλι ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 5 ονομαστική αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Vote is now closed. Πέρα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ονομαστικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9 και πάλι με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Vote Πέρας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 10. Σε δύο τμήματα, ονομαστικά, αρχίζει για το πρώτο τμήμα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. παράγραφος 11, ονομαστικά, αρχίζει τώρα. Η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14 και πάλι ονομαστικά αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 15 σε τρία τμήματα. Όλα ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Αρχίζει τώρα ψηφοφορία. Ονομαστική. Πέρας. Και εγκρίνεται και το τρίτο. Παράγραφος 16. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 8. Ψήφι υπέρ κατά αποχές. Θα χρειαστεί έλεγχος παρακαλώ γι' αυτό, για το 8. Μπορούμε να ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται, σαφέστατα. Αιτιολογική σκέψη C ε, σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ε, ε, ε, H υπέρ ε, συγγνώμη, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη H σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο, υπέρ, κατά αποχές θα το ελέγξουμε αυτό το δεύτερο τμήμα της αιτιολογικής σκέψης H. Πέρασε. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Ι υπέρ κατά αποχές. Ας το ξαναπροσπαθήσουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη και με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, πι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Q σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, θεολογική σκέψη τι σε δύο τμήματα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. X, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Α1, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. να ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ψήφιπε Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Ο εισηγητής ε, ήθελε και πάλι το λόγο. Ναι, επειδή η ψηφοφορία είχε αυτή την έκβαση, άλλαξε την έκθεση και ε, την αλλίωσε και θα παρακαλούσα να αποσύρετε το όνομά μου. Την παραδίδω. Thank you. Your request has been... Uh, Μάλιστα, το έτοιμά σας σημειώνεται. Και προχωρούμε στην επόμενη ψηφοφορία έκθεση της κυρίας Ναντέλτσεβα. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ε, παράγραφος 20 ψήφι υπέρ. Παρακαλώ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Σε δύο τμήματα ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 ε, υπέρ κατά το δεύτερο τμήμα μάλλον κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 23 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 27 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 28 υπέρ Θέλετε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 27. Μάλιστα, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε όντως. Παράγραφος 28. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 30. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτό θα ήθελα να το ελέγξουμε παρακαλώ. Παράγραφος 31. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Το δεύτερο τμήμα της 34 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρασα. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 45 ψήφι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφο 48 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 52 σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχο στο ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα της 52. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, το τρίτο τμήμα τώρα της 52. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 53 και πάλι σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές ε, ήταν οριακό, παρακαλώ να το ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα της 53. Πέρας. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα, ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 55 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, όχι και πάλι ήταν οριακό να το ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα της 55. Τώρα κλείνει η ψηφοφορία εγκρίθηκε. 58 σε τρία τμήματα, τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, το τρίτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η παράγραφος 60 σε τρία τμήματα, τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ, κατά αποχές στο ε, ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 60 πέρας δεν το τρίτο τμήμα της 60 ψήφι πέ κατά αποχές εγκρίνεται 61 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 61 πέρας εγκρίνεται παράγραφος 65 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 66. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ προφορική τροπολογία του κυρίου Σιλβέστρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην παράγραφο 66 μετά τη φράση που λέει ότι επιμένει στο γεγονό ότι οι γυναίκε ε, πρέπει να έχουν ε, δικαίωμα στο να αποφασίσουν μόνες του ε, για την αναπαραγωγή, για την αντισύλληψη και για την άμβλωση. Εγώ προτείνω το εξή μετά την άμβλωση. Αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα στη ζωή του εμβρίου. Η Κομισιόν λοιπόν καλείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να στηρίξει την εγκυμοσύνη εφαρμόζοντα τι κατάλληλε πολιτικέ. που θα επιτρέπουν στη γυναίκα όπου είναι αυτό απαραίτητο ε, να μην καταφεύγουν στην άμβλωση. Αυτό είναι μια ε, προφορική τροπολογία έτσι ώστε που δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα να ε, αποφασίζει μόνη της έτσι ώστε να μην αγκασμένη να καταφεύγει στην άμβλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Διαφωνεί κανεί με αυτή την προφορική τροπολογία. Από ό,τι φαίνεται σαφέστατα διαφωνούν, συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Δεν θα ε, ψηφιστεί λοιπόν η προφορική τροπολογία. Επανερχόμαστε στην παράγραφο 66 ως έχει σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονική επαλήθευση του πρώτου τμήματος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε and that is adopted. The... Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα ψήφι Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Ε, για το δεύτερο τμήμα ελέγχουμε έτσι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και το τρίτο τμήμα ψήφι Those against κατά αποχές εγκρίνεται. Αν θέλετε έλεγχο, εντάξει, για το τρίτο τμήμα άρχεται η παλήθευση λοιπόν, 66-3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 76. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και το σχέδιο ψηφίσματος στο σύνολό του ψηφίπε κατά, αποχές. Νομίζω ότι θα χρειαστεί επαλήθευση εδώ. Παρακαλώ ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε την τελική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Αγκρίθηκε. Η, τελευταία μάλλον έκθεση για σήμερα είναι η έκθεση κυρίας Πλάν για τη γυναικεία φτώχεια. Ψηφίζουμε την παράγραφο 8 με χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15 ψήφι υπέρ κατά αποχές αυτό θέλει έλεγχο. Ελέγχουμε την παράγραφο 15 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας. Mm. Απορρίπτεται. Η παράγραφος 16 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές θα το ελέγξουμε αυτό. Το δεύτερο τμήμα της 16 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα χρηστεί έλεγχο αυτό γιατί 34 παρακαλώ. Παλήθευση. Vote is now closed. Πέρας. Έχει σαφώ απορριφθεί. Παράγραφος 38 σε τέσσερα τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα Τσεκ! Εντάξει, το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 38 ελέγχουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το τέταρτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η παράγραφο 43. Σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 43 ηλεκτρονική επαλήθευση του τρίτου τμήματος. πέρα. Εγκρίνεται. Παράγραφο 44, ψήφι κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η παράγραφος 45 σε τρία τμήματα, τμήμα πρώτο ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές Το τρίτο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 48 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 49. Ψήφι Π. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 50. Κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ψήφι Π. Δεύτερο τμήμα. Συγγνώμη, πρόεδρο. I'm sorry. I'm... Ζητώ συγγνώμη, έχω κουραστεί. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε κουραστεί. Λοιπόν, Παράγραφος 50, τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 56, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 59 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 60 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. 62 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 65 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. 69 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. Η 77 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Παράγραφος 84. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ετυλογική σκέψη ή υπέρ. Κατά. Έψιλον ε, δηλαδή. απορρίπτεται. Εν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το σύνολο του ψηφίσματος ψήφιπε κατά αποχές εγκρίνεται. we now come... Και τώρα ερχόμαστε στις ευεξηγήσεις ψήφου. Angelis on the Schademoser report.